Okay, colleagues, um... Αγαπητοί συνάδελφοι, με τις ψηφοφορίες. Κοινή συνεδρίαση με τη Γιούρη. Ο κύριος Καβαντά, αντιπρόεδρος της Γιούρη, θα μας κάνει την ε, ανάγνωση για το κομμάτι που αφορά τη ΛΥΜΠΕ. Ξέρετε ότι έχουμε συμφωνία για το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη μετά τον πολιτικό διάλογο της 10ης Μαρτίου. Υπάρχει επιστολή του Συμβουλίου που καταγράφει την ε, πρόοδο της 19ης Μαρτίου και των θέσεων αντίστοιχα του Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου με συνένεση ότι έχουν συμφωνήσει και προχωρούν ε, τα δύο όργανα και έτσι το Συμβούλιο την 1η Απριλίου ανταποκρίνεται στην επιστολή του κυρίου Ταγιάννη. Ξέρω ότι δεν τρελαίνεστε με αυτά που ακούτε, δεν σας συναρπάζουν φοβερά. Αλλά, βάση περιπτώσει, περιγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος. Όχι, εντάξει, να μιλάτε άμα θέλετε. Ξέρω ότι δεν είναι και τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέω, αλλά όταν μιλάει ο κύριο Καβαντάκη, όταν έρθει η ψηφοφορία, παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Ψηφοφορία λοιπόν με μία ψήφο, άρθρο 55 του ιστορικού κανονισμού και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γιούρη, Ζωμαρή Καβαντά, παρακαλώ. Κύριος Καβαντά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν συνηθίζω να ενοχλώ αυτού που έχουν άλλε δραστηριότητε, αλότερε δραστηριότητε, Απλώ παρακαλώ να τι αναπτύσσουν εκτός τη αιθούση, γιατί δεν είμαι τόσο ευγενικό όρο, Κλοντ. Ευχαριστώ καταρχά αγαπητέ Κλοντ, την επιτροπή σα, Ο κύριο Φόποντα, τη συγγνώμη που δεν είναι εδώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στην ουσία του κειμένου, στα όσα είπε ο κύριος Μωράης. Απλώς, εδώ βλέπετε για τελευταία φορά έναν συνάδελφό σας που ζει ένα, μια τραγωδία, χωρίς να θέλω να μιλώ δημαγωγικά, ε, το οποίο λοιπόν η χώρα αντιμετωπίζει μια τραγωδία άνευ προηγουμένου και μπορώ να την παρομοιάσω με αυτούς που αγοράζουν ένα τουφέκι για να αυτοπυρποληθούν στα πόδια. Με όλη την ε, συμπάθεια που τρέφω για τον Κλοντ και τη συνεργασία, χάρη και στη συνεργασία που είχαμε με τον ε, Κλοντ στην Επιτροπή σας, ε, τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση για τον ίδιο και τους συναδέλφους του. Και έτσι με ιδιαίτερη χαρά συμπροεδρεύω μαζί του. Αγαπητοί φίλοι, παρακαλώ. Κύριε Μωρές, νομίζω ότι μπερδεύτηκαν οι συνάδελφοι. Πάντως το ζώμα Μαγί τον γνωρίζω εδώ και χρόνια και ήταν πολύ ευγενικά τα λόγια. Σου ευχαριστώ. Εμεί στη Λίμπε δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια αυροφροσύνες. Και που μας τα και σε τόσο ωραία γαλλικά, με τον ευγενικό σου τρόπο. Είναι συνηθισμένοι να μιλάνε, συνάδελφοι, την ώρα που μιλάω κι εγώ. <laughs> Ναι, μα γι' αυτό και προσπαθώ να λάβω από... Απέφυγα μάλλον να προεδρεύσω τη ΛΥΒΕ από το 2009, γιατί δεν ε, προτιμώ να βρίσκομαι σε δυσάρεστη θέση ποτέ, ποτέ, τις αποφεύγω πάντα. Ε, η κυρία Χάουταλα, στη συγγνώμη, δεν θα έρθει σήμερα. Η κυρία Ρέντα, αν δεν απατώ με την εκπροσωπή, εάν είναι εδώ. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω την ιδιαίτερη μου χαρά που έχω να της δώσω το λόγο. Κυρία Ρέντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. κυρία Χάουταλα, στη συγγνώμη, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις Αναφερόμενοι προς επιτροπές, ε, Γιούρι και Λίμπη είχε υπογραμμίσει την υποστήριξή της ε, προς το κείμενο καλεί όλους τους ε, συναδέλφους να το υπερψηφίσουν. Κύριο επίτευγμα του Κοινοβουλίου μας λέει είναι ότι υπάρχει το νέο άρθρο 3α για το mainstreaming. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου επίσης προβλέπεται στους δείκτες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος. Η ανεξαρτησία δε και η ουδετερότητα τη δικαστική εξουσία, ο σεβασμό του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων υπογραμμίζονται και περιγράφονται πολύ καλύτερα στου στόχου του προγράμματο. Το κράτο δικαίου και οι ευρωπαϊκέ αξίε είναι αντικείμενο όλων των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, όχι μόνο αυτών που αφορούν αξίε και δικαιώματα. Ε, ωστόσο, χρειάστηκε να γίνει σχετική προσαρμογή του προγράμματο. Το κείμενο που ψηφίζουμε σήμερα είναι μερική συμφωνία μια κοινή συνεννόηση, μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου έχει κρατήσει εντό παρενθέσεως ορισμένα σημεία για τα κομμάτια εκείνα που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει, οι οποίε θα συνεχιστούν στην προσεχή θητεία. Η κυρία Χάουτελ έχει ζητήσει από τι επιτροπέ μα να μην ψηφίσουν, είχε ζητήσει να μην ψηφίσουν πριν από το Συμβούλιο, πριν το Συμβούλιο δηλαδή να διατυπώσει σαφώς τη γνώμη του, όπω έχει εντωμεταξύ πράξη σήμερα απαντά στη διάσκεψη των Πρόεδρων και την επιστολή της, το Συμβούλιο για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, περιγράφοντας τη συμφωνία και το, προσ... το προσαρτημένο κείμενο. Η κυρία Χαουτέρα λοιπόν λέει ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιντενχελτσερ ε, από τη Λίμπε, σκιώδης δεν είναι εδώ. Μπυρκίτα Ζίπλ, έτσι δεν είναι. Κυρία Ζίπλ, δεν έχω τίποτα να προσθέσω στα όσα είπε η κυρία Ρέντα. Πολύ ευχαριστώ να γίνει η ψηφοφορία σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Καλώ ψηφίζουμε λοιπόν. Με μία ψήφο. Ηλεκτρονικά. Αν έχετε όλες τις κάρτες μαζί σα. Θα καταγραφεί η ψήφο σας παρακαλώ. Αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 49 υπέρ 7 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής και τους Κιώδης αλλά και τους ε, συναδέλφους της Γιούρη. Και τώρα μπορούν να μείνουν ε, τα μέλη της ΛΥΜΠΕ μόνο για να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ, Ζωμαρή.